Hello everyone, good morning. σε όλους σας. Θα ήθελα να προετοιμάσετε τις ε, κάρτες σας για την ε, ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. First of all, I want to welcome uh, Madam Dana Balkarova, Chair of the Committee of Ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την κυρία Μπαλκάροβα, πρόεδρο του Περιβάλλοντο του ε, Κοινοβουλίου τη Τσεχική Δημοκρατία. Σα καλωσορίζουμε, κυρία Μπαλκάροβα. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ε, έκθεση φορά την αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού ανώτατα όρια καταλήπων για την ουσία ασεταμιπρίντ σε ορισμένα προϊόντα. Και θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. The next one. Η επόμενη έκθεση αφορά την προφορική ερώτηση καταστρατήγηση του, καταστρατηγήσεις του Natura 2000. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την ίδια ε, προφορική ε, απάντηση, αλλά προς το Συμβούλιο, ερώτηση, συγγνώμη, στο Συμβούλιο αρχίζει αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Now we are voting. Συνεχίζουμε. για το σχέδιο γνωμοδότηση προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη τη Γενέβη Συμφωνία τη Λισαβόνα για τι ονομασίε προέλευση και τι γεωγραφικέ ενδείξει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης. Τώρα ψηφίζουμε. για τις ενέργειες, τροπολογίες της Ενέργειας Ένωσης μετά την προσχώρηση στην πράξη της Γενέβης Συμφωνίας Λισαβόνας της Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικές ενδείξεις. Υπάρχουν πολλές ψηφοφορίες οι οποίες είναι διατύπωσης και γλωσσικές που κατέθεσε ο κύριος Φλάνεγκ. Και δεν θα περάσουμε στις λεπτομέρειες που αφορούν αυτές τις ε, γλωσσικού περιεχομένου και διατύπωσης τροπολογίες. Δεν θα τις ψηφίσουμε. Αναφέρεστε στη γραμματεία και κάνει τις γλωσσικές διορθώσεις. Τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αριθμός 1, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ΕΛΚ ήταν υπέρ. Άρα απορρίπτεται ή θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Να επαναλαμβάνουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Βασικά, εγκρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. Επόμενο θέμα. Εδώ, εδώ είναι το μεγάλο θέμα μας. Λοιπόν, διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κυρία Ζάμερ. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεση. Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 ε, με συγχωρείτε. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα τη και εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 5. Συμβεστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 229. Διανάταση ισχυρός 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 230. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.32, 2.33 και 2.34. Όχι, είναι διαφορετική. 2.32, 2.33. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 2.34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά 269 σελίδα 15 η 268 ε, γράφει πάνω no vote ψηφίζουμε λοιπόν τη 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 269 I've seen that coming. Το περίμενα. Πέρας ψηφοφορίας. Κυρία Μάκε, είστε υπέρ χωρίς κάρτα, οπότε εγκρίνεται. 2,70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,72 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 286 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 288 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζική ψηφοφορία 1 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε block vote 1. The vote Πέρα στις ε, η κυρία Γατημάκη απέχει, οπότε απορρίπτεται και κάποιος δεν ψήφισε. Block vote 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να δούμε την 2. Ας ψηφίσουν όλοι αυτή τη φορά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξεκολουθεί κάποιος να μην ψηφίζει. Τώρα ψηφίζει. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 290 292 συγγνώμη 290 2,90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 πια μου λένε ότι 26 είναι στο block vote 2. 28 συγγνώμη είναι στο block vote 2. 2.93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 2.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι βέβαιο. 2.96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ «29 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 2.97 Άρχεται η ψηφοφορία για τη 297. Η κυρία Γιατεμάκη είναι υπέρ. «2.97 δεν θέλουν να ψηφίσουν όλοι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη, γιατί η κυρία Γιατεμάκη ήταν υπέρ. όταν σκέφτομαι τις ε, ψηφοφορίες αν μπλοκ σε αυτό το αίθουσα ε, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη αν κάποιος δεν θελήσει να ψηφίσει πρέπει το αποτέλεσμα 2,98 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 2,99 εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία από τους πράσινους είναι όλοι κατά είναι κανείς κατά της προφορικής αυτής τροπολογίας όχι να ψηφίσουμε την 299 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 300 όχι. Τζούρι 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 τμήμα 2. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Άλντε. Τι κάνατε για αυτό. 307 τμήμα 2. Είστε κατά, ε. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και η κυρία Γιατεμάκη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τζουρί 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.13 έχουμε μια προφορική τροπολογία που ζήτησε η Γκουε. Είναι κανείς ε, κατά. Ναι, κυρία Ζόμερ, είστε κατά. Πρέπει να πείστε άλλους πέντε ανθρώπους. 13 ψηφίζουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3-15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3-17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3-18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 328 για τις άλλες δύο δεν έχουμε ψηφοφορία 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 328 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Η κυρία Γιατεμάκη έχει την κάρτα της πλέον. Εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 332 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «3.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ Ήταν πολύ καθαρό, αλλά να το ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την 333. Τι είπα, απορρίφθηκε. Εγκρίνεται. Διότι το ΕΛΚ ψήφισε επίση το ίδιο. Ευχαριστώ. Πάω λίγο πολύ γρήγορα. Η συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Δεν ψηφίζουμε την 37. Συγγνώμη. 3.39 και 3.40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Εγκρίνεται. 3.38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, μπέρδεμα λίγο στο Άλντε. Ε, το ΕΛΚ είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ίσως να κάνουμε ε, κατά τμήματα ψηφοφορία. Όχι, πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα 3, 42, 43, 44 και 45, οι οποίε είναι ταυτόσιμε. Άρχεται ψηφοφορία. Συγγνώμη να δω. Με ανάθεση χειρό υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτονται, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Was adopted? Yeah. 347 mm-hmm. then. Who is in favor? Against. 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 350 υπέρ κατά αποχές Να ελέγξουμε την 350. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούρι 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 353 και η Γιούρι 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ 350 λάθος 358 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 360 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε 360 άρχεται η ψηφοφορία και πολύ μικρό α, πέρας απορρίπτεται 361 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 361 Πέρας. Απορρίπτεται. 362 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Closed. Adopted. Πέρασε, εγκρίνεται. Which one? No, she's talking to Peter. Ah, I'm sorry. <laughs> I thought I jumped over something. Ζητώ συγγνώμη, νομίζω ότι παρέψα κάτι, νόμιζα, αλλά... Δεν εγκρίθηκε η 366. 366. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. <clears throat> Θέλω να πω ότι εγκρίθηκε, θα ήθελα να ελπίζω, αλλά... Εγκρίνεται. 67, who is in favor. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 368 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται Γιούρι 72 υπέρ κατά αποχή Άλτε είναι υπέρ εγκρίνεται να ελέγξουμε Vote closed. Ah, rejected. Πέρας προφορίας, απορρίπτεται. 369, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 73 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε The vote is closed. Adopted περσοφορίας εγκρίνεται. 371 372. 371 και 372 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 373, 374 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. 375 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Αποχές. Παρακαλώ να επαληθεύσουμε. Πέρας. Απερίφθη. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 384 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Επαλήθευση λοιπόν. Πέρας, απερίφθη. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 390 και 91 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζούρι 70 όχι, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. 3,94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3,95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 399 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Φαίνεται πως πρόκειται για σφάλμα στην ε, λίστα ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τότε block vote όλες μαζί, δηλαδή τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται επαλήθευση, επαλήθευση. Πέρας, εγκρίνεται ή μάλλον εγκρίνονται τώρα. Τζούρι 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεν ακολουθούν, μάλλον δεν υπάρχουν άλλες ψηφοφορίες. 403 και 79 τζούρι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 404 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 405 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 410 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 414 υπέρ. Κατά. 414 υπέρ, λέει η πρόεδρος πάλι, 414 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 415 υπέρ, επαλήθευση για την 414. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία 31-29. Α, όπως βλέπετε, είχα δίκιο. Ε, σας το είπα ακριβώς. Ωραία, 415 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζούρι, 82 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 416 και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τζούρι 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πες 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζούρι 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούριο 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τζούριο 85. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 89 υπέρ. Κατά. Αλτε είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Νομίζω λοιπόν ότι εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Ενεκρίθηκε. Ναι, 4.40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 441 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4.42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 443, 44 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 446 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 447 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 450 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 452 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Αρχίζει. Και τέλος. Ενεκρίθη. 53. Α, λέει no vote. Block vote 1 και 2, 1 και 2 εγκρίθηκε, αλλά τούτη εδώ δεν εγκρίθηκε. Ε, λέει κάποιος χωρίς να γνωρίζουμε ποια φωνή ήταν αυτή. Τώρα, πρόεδρος, μου λένε ότι αυτό αποτελεί μέρος, αυτή εδώ αποτελεί μέρος της Block Vote 2 και αφού απερίφθη η Block Vote 2 σημαίνει ότι καταπίπτει και η 53. Αν όμως θέλετε να το αλλάξετε, η κυρία Κάντενμπαχ επίσης λέει ότι είναι τμήμα του Block, του συνόλου δηλαδή των τροπολογιών φαίνεται πως 53 και Jury 91 ταυτίζονται, ώστε καταπίπτουν αμφότερες. Καλώς. Μίλαγα λίγο και στον εαυτό μου, λέει η πρόεδρος, να με συγχωρείτε. Ωραία λοιπόν. Jury 91 και 53 είναι ταυτόσιμες και συναποτελούν μέρος του Block Vote 2. Γι' αυτό και δεν ψηφίζω πλέον, διότι απερίφθησαν όλες μαζί αυτές. Άρα τώρα 452. Α, την ψηφίσαμε, ωραία, και εγκρίθηκε. Τζούρι 92, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 355 και 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 457 και τζούρι 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 458 και 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 460 και 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 464 και τζούρι 95. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 465 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 55 τώρα. Α, με συγχωρείτε, 467 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καλώ λοιπόν, τότε α ψηφίσουμε την 467, ηλεκτρονικά εννοώ. Πέρας, απερίφθη. 468 και 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 470 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 471 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Τζούρι 97 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τζούρι 98 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 473 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 475 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 476 και τζούρι 101 λέει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές είναι κάπως ε, ασαφές το αποτέλεσμα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτό είναι το δικό μου. 477 και τζούρι 101. Εγκρίνονται λοιπόν. Πηγαίνετε στην τζούρι 102. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 478 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 479 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 483 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 483 αρχίζει. Πέρας. Και ενεκρίθη. «484 υπέρ». Κατά αποχές απορρίπτεται. 486 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 487 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 488 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 489 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 491 και 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 493 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 494 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 495 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 496 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 497 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τζούρι 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 499 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 501 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 107 υπέρ. Κατά αποχές. Τσεκ. Επαλήθευση. Είστε κατά εσείς οι πράσινοι. Α, απέχετε. Καλώς. Λοιπόν, αρχίζει, τώρα τελειώνει. Απερίφθη λοιπόν. Αλλαγή πλέον στις ισορροπίες. Ε, συγγνώμη, 502 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 503 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 504 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 505 και 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 507 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 508 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 509 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 510 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 511 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 513 και 14 υπέρ κατά επαλήθευση. Τέλος, ενεκρίθη. 510, όχι αυτή ενεκρίθη, 515, 521 στην επόμενη σελίδα στο έγγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τέλος. Απερίφθη. 522 και τζούρι 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 524 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Πάμε ότι δεν ήταν τόσο σαφές. Πέρας. Εγκρίθηκε. Κάπου εδώ δεν ε, με ξεγέλασε η ECR. Λέει η πρόεδρος. 526 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 529 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 530 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 532 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 534 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 535 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 536 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά κάνω επαλήθευση Πέρας. Εγκρίθηκε 31-28. Τζούρι 110 και 537 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 538 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 539 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές επαναλαμβάνω 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά θέλετε επαλήθευση για την 64 καλώς επαλήθευση πέρας εγκρίθηκε. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τζούρι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τζούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά η πράσινη Ας επαληθεύσουμε την 73. Ε, Πέρασε και εγκρίθηκε. Πού βρισκόμαστε ακριβώς. Τζούρι 3. Ωραία λοιπόν. Η ψήφη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τζούρι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τζούρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τζούρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλίας 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 και τζούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Στη... Ε, γεια σας λέει η πρόεδρος σε κάποιον που φταρνίστηκε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Τζούρι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 111 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μα είναι και σοσιαλδημοκράτες και λαϊκό κόμμα αντίθετοι στην ψηφοφορία. 112 υπέρ. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τζούρι 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. 18 ε, τώρα τζουρί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 και τζούρι 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τζούρι 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τζούρι 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Υπαριθμόν 11 υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 153 και τζούρι 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μια στιγμή. Σοσιαλδημοκράτες και, Λαϊκό Κόμμα κατεψήφισαν. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αλλά σε επαληθεύσουμε. Δεν ήταν σαφές το μήνυμα των χειριών. Τελειώνει πια η ψηφοφορία σιγά σιγά. Πέρας. Απερίφθη. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 29 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ας το ξανακάνουμε. 164 υπέρ. Ε, είναι κρίση γιατί βλέπω καθαρά από τα χέρια. Τώρα, τζούρι 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τζούρι 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, θέλετε επαλήθευση. Επαλήθευση Τζούρι 34. Όπως η μόνη που κατεψήφισαν ήταν του Λαϊκού Κόμματος νομίζω. Θα το δούμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία Ορίστε, θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Χόισλινγκ. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πριν από την τελική ψηφοφορία. αν συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες. Λίγα λεπτά. Δύο λεπτά σας δίνω, λέει η πρόεδρο. Δύο λεπτά. Α του δώσουμε δύο λεπτά. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν ακόμη. Δύο λεπτά. Which is the next one? This one. Supplementary protection certificate, which is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 Final vote. Everyone is, uh, Η πρόεδρος. Είστε όλοι έτοιμες και έτοιμοι να ψηφίσετε. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Τέλος. Εγκρίθηκε. Now we are voting on... Uh, Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία, για διαγνωμοδότηση για τα πιστοποιητικά συμπληρωματική προστασία για ιατρικά προϊόντα. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 4. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 7. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 10. Συμβιβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.29 και 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2.31, 2.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ Ποιος είναι υπέρ της 23 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 και 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 35. 35. Τροπολογία 35. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά υπενθύνεται. 13 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise 15. In favor, again. Εγκρίθηκε η συμβαστική 15. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ίσως, ας κάνουμε όμως ηλεκτρονική επαλήθευση της 88. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται όντω. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Έχουμε δύο τροπολογίες, την 118 τώρα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και την 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση.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 αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 76 αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση? Όχι. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 81 ήταν αυτή. Ηλεκτρονική επαλήθευση. And it's Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 87. Κύριε Πεντιτσίνη, δεν είναι δική σας η τροπολογία. Τέλος πάντων, αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ηλεκτρονική επαρήθευση. Απορρίπτεται. 87. Ναι, ναι, έχετε τέσσερις πολιτικές ομάδες που ψηφίζουν ε, κατά, εν πάση περιπτώσει. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 108. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 109. Απέχει η Άλντα. Λοιπόν, α κάνουμε επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 114, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 116. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 και 121 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση λίγη ψηφοφορία εγκρίνονται 120 120 υπέρ κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές 141 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. διότι ψήφισαν χωριστά κάποιες ομάδες. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 146 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά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 κατά, αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, ε, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 και 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, Εισαπορρίπτεται. 15. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά, 16 και πάλι επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Η 20 είχε αποσυρθεί. Αυτό έχω εγώ στον κατάλογο. Ίσως δεν το έχετε εσείς μπροστά σας. Γι' αυτό το Πήγα στο 21 και τώρα είμαστε στην ψήφιση της 22. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Now we are voting on Πάμε να ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες ε, για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Πάμε λοιπόν. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ, ε, ψηφοφορία unblock, 29, 36 και 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να το ελέγξουμε ξανά 31 υπέρ κατά απορρίπτεται 32 υπέρ εντάξει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 31 31 ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας Παραδέχομαι, είχα τύχει, αλλά απορρίπτεται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θεώρησα ότι οι πράσινοι θα υποστήριζαν το ΕΛΚ. 99,9 των περιπτώσεων της 100 των περιπτώσεων 32. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται on block μέχρι την 46 συμφωνείτε 37 έως και 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα unblock 48 έως 60 και 61. Ε, μέχρι 60, 48 με 60, ποιος είναι υπέρ. Εσείς πείτε μου κύριε Πεντιτσίνη. Okay, 48 to 51. 48 με 51, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κύριε Πεδίτσινη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Unblock τώρα. 53 έως 60. 53 έως 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Unblock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 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές. 8 υπέρ είναι και ποιος υπέρ της 8. Α, αλλάζω τα πράγματα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 11. Και το άλλο δεν είναι υπέρ. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται παρόλα αυτά. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία And it closed. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας με τις ψηφοφορίες. Εδώ ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες και έχουμε την εκδήλωση με, τους, με την νεολαία στις 11. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα για καφέ, αλλά παρακαλώ να είστε πίσω για την εκδήλωση I. Ναι. Καλό θα ήταν να είστε εδώ, θα τα πούμε στις 11.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

τεστ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 Well, Καλώς ήρθατε όλες και όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά δεχόμαστε σήμερα τρεις εκπροσώπους της νεολαίας που ήρθαν στο European Youth Event στο Στρασβούργο τον Ιούνιο που μας πέρασε. Ε, η φετινή ας πούμε έκδοση αυτού του αναδιετία τελούμενου ε, γεγονότος έχουν ε, με συμμετοχή πολλών χιλιάδων νέων και των δύο φίλων και το Προεδρείο αποφάσισε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές η έκβαση δηλαδή της προσπάθειας αυτής με ακρόαση ώστε να υπάρξει διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των νέων αμφωτέρων των φίλων ε, ε της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους τις οποίες θα ακούσουμε. Έτσι λοιπόν μετά από την τρίτη ε, έκδοση του ΆΙ έχουμε τρία πρόσωπα, τρεις νεαρές ε, ε, κοπέλες οι οποίες θα μας αναπτύξουν τις ιδέες τους. Η κυρία Βίβιαν Μπέργκερ για θέματα δημόσιας υγείας, η κυρία Πράντινες για θέματα ε, αποβλήτων και τέλος η κυρία Αναμαρία Ρένερ που θα μιλήσει για βιώσιμη διαβίωση νέοι και νέε από όλη την Ευρώπη μας παρακολουθούν τώρα στο web stream, δηλαδή μέσω του διαδικτύου, μπορούν να μας παρακολουθήσουν και από τα κοινωνικά μέσα, από το Twitter, είτε και από τι οθόνε και μπορούν να ε, στείλουν και tweet με το σχετικό hashtag, το οποίο ε, το βλέπετε και στην οθόνη. hashtag i2018, δηλαδή 2018 ε, ε, ε, Σε παρεμβάσει των δύο λεπτών θα έχουν την ευκαιρία οι ευρωβουλευτές να απαντήσουν ή να τοποθετηθούν. Και τώρα για το ζήτημα της υγείας. Της υγείας. Οι νέοι μίλησαν για τη μαζική χρήση των κοινωνικών μέσων και την επίπτωση στην υγεία για το ηλεκτρονικό ιστορικό των ασθενών, για θέματα παχυσαργίας των παιδιών. Κυρία Γκέργερ, σας δίνουμε ε, τώρα τον λόγο για το European Electronic, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ελεκτρονικό Ιστορικό των Ασθενών. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάζω την ιδέα ενός τυποποιημένου ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από επαγγελματίες και από τους ασθενείς. Ε, πρόκειται για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικά αποθηκευμένων ε, πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή επιπλέον. Η μελέτη των επιδημιολογικών ε, πληροφοριών του πληθυσμού μπορεί να μελετηθεί μέσω ενός τέτοιου εργαλείου. Στο έκτο έτος ιατρικής όπου σπουδάζω έχω ζήσει τις δυσκολίες ε, του ιατρικού προσωπικού με τα πολλά αρχεία και τα διάφορα ε, υπολογιστικά συστήματα και τις διαφορετικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Σημαντικές πληροφορίες χάνονται, συνταγογραφούνται ε, φάρμακα με λάθος τρόπο και μερικές φορές τα λάθη είναι μοιραία. Οι πληροφορίες των ασθενών λοιπόν θα αποθηκεύονται σε ένα φορητό σύστημα όπως μια κάρτα και τα στοιχεία θα ενημερώνονται διαρκώς από τους επαγγελματίες και από τον ασθενή με μία επίσημη εφαρμογή θα μπορεί ο ασθενή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ανα πάσα στιγμή και να ενημερώνει του ε, ιατρικού επαγγελματίε ανα πάσα στιγμή, για παράδειγμα όσον αφορά τι τιμέ του ζαχάρου, με διάφορε προειδοποιήσει που θα βοηθούν στην καλή κατάσταση του ασθενή και στην κατανόηση ορισμένων θεμάτων υγεία. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ένα τέτοιο αρχείο πρώτα σε εθνικό επίπεδο και μετά σε όλη την Ευρώπη. Πρώτον, πολλά ηλεκτρονικά αρχεία κυκλοφορούν από διαφόρους παρόχους ήδη στην αγορά. Με... Τα προϊόντα είναι πολλά και διαφορετικά, ωστόσο είναι πολλές και διαφορετικές και οι ποιότητες ε, και ο χειρισμός των δεδομένων. Βρίσκονται ακόμα σε ανώριμο στάδιο ένα επίσημο ευρωπαϊκό ιατρικό αρχείο μπορεί να συγκεντρώσει σε ένα σύστημα όλα τα στοιχεία αυτά για όλους τους ασθενείς. Η επιδημιολογική αξιολόγηση ανώνυμων δεδομένων ασθενών είναι μια άλλη δυνατότητα που παρέχουν τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και που θα πληρούν και τις, και, ε, τις προϋποθέσεις του GDPR. Πρόκειται για μια πρόοδο πολλά υποσχόμενη και η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα πρέπει να επενδύσει σε αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε τώρα να μας μιλήσετε για την παχυσαρκία και μετά θα ακούσουμε τη ε, σχόλια για το όλο θέμα. Η δεύτερη μου ιδέα αφορά την παχυσαρκία. Σύμφωνα με τον Παγκοσμίο Οργανισμό Υγείας το 2008 το 50% ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, υπερβαροί και 20% παχύσαρκη ο συνδυασμό υπερβολική διατροφή, ε, έλλειψης άσκησης ε, και γενετική ε, έχει κάνει την παξαρκία παγκόσμια επιδημία. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από πολλές οπτικέ γωνίες. Το πρώτο μέτρο που θέλω να προτείνω αφορά την έλλειψη άσκησης. Ένα τρίτο των ενηλίκων στην Ευρώπη δεν ασκούνται επαρκώς σωματικά. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να προσφέρει λοιπόν δύο ώρες αθλητισμό στους υπαλλήλου τη ε, κάθε εβδομάδα. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο πολλών θανατηφόρων ε, μη μεταδοτικών ασθενειών. Προτείνω τρία σημεία στα οποία μπορεί να δράσει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γυμναστήρια, ντου και εξοπλισμού στι εταιρείε ε, με βοήθεια οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στούντιο, πισίνες επίσης με επιχορήγηση και ε, συνήθειες όπως η γυμναστική και η γιόγκα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ε, στις εταιρείε μέσω μιας εθνικής εκστρατείας. Το πρόβλημα της κακής διατροφής, ε, του junk food, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα ειδικό φόρο για προϊόντα με υπερβολική περιεκτικότητα στη σάχαρη. Θα πρέπει να, περι... να επισημένονται τα σχετικά προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική επιτροπή χρησιμοποιώντας το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη τα ε, προϊόντα με κόκκινη σήμανση θα πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγήσεις ώστε να επισημαίνονται τα ανθιγεινά τρόφιμα και οι ανθυγιεινές συνήθειες στον πληθυσμό. Θα πρέπει να υπάρχουν και εθνικές εκστρατείε και διαφήμιση προς ενημέρωση των καταναλωτών. Όχι ο καταναλωτής αλλά ο, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υφίσταται τον φόρο και αυτό θα αποτελεί κίνητρο για να μειώνει την περιεκτικότητα σε ζάχαρα στα σχετικά προϊόντα αυτός ο φόρος θα πρέπει να επενδύεται για συγκεκριμένο σκοπό σε ταμεία υγείας. Γιατί λοιπόν ε, όχι κεντρικό πρόγραμμα, επειδή είναι παγκόσμια επιδημία και προ... ένας, μια αιτία θανάτου που μπορεί να προληφθεί, ε, σας καλώ να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Βίβιαν. Μιλήσατε για το ηλεκτρονικό μητρό ασθενών για ζητήματα παχυσαρκίας, για επιδότηση ασκήσεων, για την παρακολούθηση του ζάχαρου στο αίμα, για ένα ταμείο υγείας. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα προσκαλέσω τους ε, συναδέλφους μου να τοποθετηθούν τώρα και πρώτος ο κύριος Βέλκεν. Μόλις τώρα έστελνα tweet σχετικά με, το, ε, με την εκδήλωση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τις ιδέες που υποβάλλετε. Θα ήθελα πρώτα να μιλήσω για το ηλεκτρονικό ιστορικό υγείας, ε, αρχείο δηλαδή, που είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα και χρειάζονται βέβαια και άλλα βήματα να γίνουν προ την κατεύθυνση αυτή. Προέρχομαι από χώρα μέλο όπου ακόμα οι, συνταγοί γράφουν, ε, με οι γιατροί γράφουν τις συνταγέ τους με το χέρι. Και βλέπω πραγματικά ότι, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη. Και λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά παρόλα αυτά να προχωρήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε θέματα e-health, ηλεκτρονικής υγείας, δηλαδή σε διάφορες γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις και ξαναείπα η πορεία είναι μακρά και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Ακούγοντας όμως από εσά ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα, ε, αυτή ε, την ε, πρότασή σας την εκτιμώ ιδιαίτερα, διότι όντως ασκεί κάποια πίεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φορολογία επί της ζάχαρης, δεν είμαι βέβαιο έχει συζητηθεί πολλέ φορές ε, στο Κοινοβούλιο, νομίζω. Ίσως οι συναδελφοί μπορούν να σχολιάσουν επ' αυτού περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό που τονίσατε είναι ε, στην ουσία ότι κάτι πρέπει να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και ότι χρειαζόμαστε κάπως περισσότερες ιδέες από απλώς αυτόν τον σηματοδότη, δηλαδή με κόκκινα, πράσινα, κίτρινα χρώματα πάνω στις συσκευασίες αλλά θα πρέπει να δείχνουμε πραγματικά στην επισήμανση, στις ετικέτες των προϊόντων, ποιο είναι το ποσοστό λιπαρών, ποιο είναι το ποσοστό ε, σακχάρων πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων. Έχουν συζητηθεί, είπα αυτά τα πράγματα ε, εδώ στο Κοινοβουλίο, έχουν συζητηθεί πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Για την ώρα το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα επ' αυτού. Επομένως, η ίσπραξη φόρων είναι ούτως ή άλλως η η θεσπιση και η ίσπραξη φόρων δεν είναι ζήτημα, δεν είναι ζήτημα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, είναι καθαρά κυριαρχία των χωρών μελών. Αυτές θα πρέπει να κινητοποιηθούν πρώτες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του θέματος και τις διάφορες ιδέες σας, τις οποίες εκτιμώ ιδιαίτερα. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα που είναι τα γερμανικά, επειδή μάλιστα παρακολουθούν ε, ε, Γερμανοί ε, ακροατές, θεατές μέσω των social media. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το πρώτο θέμα. Είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σας ότι δηλαδή χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρησης και πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα που να είναι δυνατόν να γίνεται η πρόσβαση δηλαδή παντού και πάντοτε. Υπάρχουν όμως σημαντικές αντιστάσεις και ειδικότερα στην Ομοσπονδιακή Γερμανία που γνωρίζω και καλύτερα ποια είναι η κατάσταση. Προσπαθήσαμε να το περιλάβουμε και στα δικαιώματα των ασθενών και αντιστάθηκαν πάρα πολύ ιδίως οι ιατροί. Η τεχνολογία αυτή δεν μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί χωρίς κανέναν έλεγχο. Ίσως έχετε συζητήσει μεταξύ σας και το ερώτημα ε, πώς μπορούν να υπερκεραστούν αυτές οι αντιστάσεις, ιδίως σε πιο ηλικιωμένους ιατρούς σημειώνονται σημαντικότατες αντιστάσεις. Οι νεαρότεροι ιατροί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα αυτά. Και εάν αναζητήσετε ίσως νεαρούς ιατρούς ή φοιτητέ της ιατρικής, ίσως να υπάρξει μια κίνηση εντονότερη. Τώρα για την φορολογία ανεξαρτήτως του πώς τοποθετείται κανείς απέναντί της, υπάρχει ένα σημαντικό κόλλημα. Ε, είπε ο Τίμο Βέλκεν ότι, που μίλησε πριν από μένα ότι ε, δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής φόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει απολύτω. Έχει δικαίωμα, αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσει το Συμβούλιο Υπουργών. Σε κάθε χώρα μέλος η υπόθεση αυτή είναι και διαφορετική συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκλογική μου περιφέρεια το θέμα της επιβολής φόρων στο καύσιμο ντίζελ. Ε, αυτά δεν βρίσκουν σε όλους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να προωθηθεί στις χώρες μέλη. Αν δηλαδή θέλει η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί, πρέπει να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη και κυρίως να ξεφύγουν από την ομοφωνία, από την υποχρέωση ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων για να περάσουν στην καταπληψηφία. λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Eichhout. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ιδέες που παρουσιάσατε και τις προτάσεις σας. Και πράγματι νομίζω πολλά από τα θέματα που αναφέρατε τα συζητούμε ήδη εδώ. Και καμιά φορά βέβαια ξεκινάει και ένας πολιτικός καυγάς, όπως πάντοτε σε πολιτικές αρένες. Η αντίσταση, όπω είπε μόλι ο Πέτερ Λίζε, προέρχεται κυρίω από τι χώρε μέλη και κυρίω ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ιστορικό των ασθενών για ηλεκτρονική ιατρική τεχνολογία. Διεξάγουμε αγώνα και εδώ στο Κοινοβουλίο, αλλά υπάρχει αντίσταση και αντίσταση και στο επίπεδο των χωρών μελών που για να καμφθεί θα είναι χρήσιμο να ασκήσετε και εσείς πίεση. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, παχυσαρκία, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ε, η πρώτη σας ιδέα για τη δημιουργία ταμείων, ε, αντιλαμβάνομαι την αξία της, έχω όμως μια αμφιβολία για το αν θα πρέπει να είναι το ταμείο αυτό ευρωπαϊκό. Δεν κυκλοφορούν και τόσα πολλά ευρωπαϊκά χρήματα από εδώ και από εκεί. Και πάλι εδώ αντιμετωπίζουμε σημαντική αντίσταση όταν καλούνται οι χώρε μέλη να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αυξήσουν τη συνεισφορά προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν είναι πράγματι και εδώ ενδιαφέρον να προωθεί η ιδέα αυτή στο εθνικό επίπεδο. Για τα φορολογικά μίλησαν προηγουμένως οι δύο συνάδελφοί μου, αλλά δεν θα με εξέπλητε εάν οι ιδέε που θα υποβάλλετε ε, συνδέονται πάντοτε με φορολογία. Είναι ένα θέμα το οποίο όντω πρέπει να συζητηθεί. Και το αυτόματο ανακλαστικό των χωρών μελών είναι να πούν «Α, μια στιγμή η φορολόγηση είναι εθνική αρμοδιότητα». Υπάρχει τρόπο να ξεπεραστεί αυτό, αλλά είναι πολιτική η συζήτηση αυτή. Διότι ακριβώ επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανή να επιτύχει αποτελέσματα στην φορολόγηση, το αποτέλεσμα τελικώ είναι ότι όλο και λιγότερο φόροι πληρώνονται, καταβάλλονται. Οι επιχειρήσεις μειώνουν διαρκώς τους φόρους που καταβάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικώς τι γίνεται, φορολογείται περισσότερο η εργασία ή μειώνονται οι δαπάνε εν τέλει. Αυτό είναι ένα θεμελιώδε πρόβλημα τη Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και χαίρομαι που θέτεται το θέμα αυτό, αλλά για την ώρα η συζήτηση αυτή θα πρέπει να μετακινηθεί μάλλον στο εθνικό επίπεδο, αν δηλαδή θα φορολογηθεί η ζάχαρη η περιοκτικότητα δηλαδή σε σάκαρο ε, διαφόρων ε, ε, καταναλώσιμων, τροφίμων ας πούμε κλπ. Τέλος, για τον σηματοδότη. Καμιά φορά πρέπει να δείξει κανείς ότι γίνεται και ένας πολιτικός αγώνας εδώ στο Κοινοβούλιο. Εμείς ως πράσινοι είμαστε πάντοτε υπέρ του σηματοδότη στις ετικέτες των τροφίμων και χάσαμε διότι αντιτάχθηκαν οι συντηρητικοί, η συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος του Κοινοβουλίου να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι η συντηρητική δεν είναι υπέρ. Α, μια στιγμή απαντά σε σχόλιο κάποιο από την ε, συντηρητική πλευρά της αίθουσα. Πρόκειται για πολιτική αρένα. Όταν εκθέτει κανείς τους πολιτικούς αυτούς αντιπάλους, αυτοί διαμαρτύρονται και δυσανασχετούν, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Και άλλα έχουν χαθεί λόγω της αντίδρασης των πρασίνων, λέει η κυρία Βάλερ. Όχι, όχι, οι φιλελεύθεροι ήταν. Τα ξέρω πολύ καλά γιατί ήμουν και σκιώδη συζητητή για το θέμα αυτό, σημείο ο κ. Σέικχαουτ. Μην δυσμονείτε ότι πρέπει να περιορίσετε σε δύο λεπτά η κυρία Κάντεμπαχ. Εγώ θα ήθελα πρώτα βέβαια να απευθύνω το θερμό καλό ορίσατε στις τρεις νέες και να επανέλθω σε αυτό που είπε ο ε, ε, κ. Σέικχαουτ για τον σηματοδότη κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα. Στην Ευρώπη έχουμε ένα από τα καλύτερα και ασφαλέστερα ε, πρότυπα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων, δηλαδή κάθε τι που καταλήγει στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ακίνδυνο για την υγεία. Βεβαίω αυτό εξαρτάται πάντοτε από τις ποσότητες, από τις δόσεις. Τώρα, εάν αναφερθούμε μονάχα στον σηματοδότη, γιατί κάθε τρόφιμο θα πρέπει να έχει ένα κόκκινο, ε, σημαδάκι, ένα κέντρο, ένα πράσινο, ένα κόκκινο θα σημαίνει ότι είναι κακό. Αλλά δεν είναι από μόνο του κακό, είναι ο συνδυασμό των συστατικών του και η ποσόστοση, η δόση που είναι κάθε συστατικό μέσα στο ε, συγκεκριμένο τρόφιμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και χαίρομαι, είμαι ιδιαίτερα υπερηφανή που τουλάχιστον για τυποποιημένα τρόφιμα και για τα σύνθετα τυποποιημένα τρόφιμα έχουμε καταφέρει να χρησιμοποιούμε αυτή τη σηματοδότηση. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε νωρίτερα, πρέπει να αρχίσουμε με εκπαίδευση των νέων δηλαδή με τον ε, αλφαβητισμό της υγείας, α το πούμε έτσι, ξεκινώντας από τα πολύ μικρά παιδιά, που όταν πίνουν ένα χυμό φρούτου, καταρχήν αυτό είναι κάτι καλό, είναι κάτι υγιές. Όμως, αν η πορτοκαλάδα έχει μέσα πολύ ζάχαρη, τότε όχι. Δεν θέλω τώρα όμως, για παράδειγμα, στην ε, φρεσκοστημένη πορτοκαλάδα να βάλω πάνω ένα κόκκινο σημαδάκι, ένα κόκκινο ετικετάκι, επειδή έχει πολύ ζάχαρη μέσα. Εδώ, ξαναλέω, χρειάζεται εκπαίδευση, διαφώτιση, ώστε να αντιληφθούν οι άνθρωποι ποια πράγματα είναι υγιή για αυτού. Ποιο είναι ο υγιεινό τρόπο διαβίωση. Παράδειγμα, περισσότερη κίνηση, περισσότερη άσκηση. Υπάρχουν πολλά σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και οι περισσότερε χώρε μέλη αντιλαμβάνονται πλέον το πρόβλημα ότι οι παιδιά και νέοι δεν κινούνται επαρκώ. Και όμω, παιδική σταθμή, νηπιαγωγία, είναι έτσι χτισμένα σε όλη την Ευρώπη, που δεν δίνουν ελευθερία κίνηση στα παιδιά. Αυτό είναι καθαρά εθνικό καθήκον να εφαρμόσουν στην πράξη δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ε, δεν υπάρχουν όμω και επαρκή ε, ευρωπαϊκά κονδύλια για να προωθήσουν τι πρωτοβουλίε αυτέ. Όταν, για παράδειγμα, συνδυάζεται και με την βελτιωμένη ενσωμάτωση. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο, άλλα ομαδικά παιχνίδια ε, συμβάλλουν πολύ και στην ενσωμάτωση στην κοινωνία των διαφόρων ομάδων. Αυτό ίσως είναι και, αυτό ίσως είναι και ένα αντίβαρο. Και βεβαίω και το έξτρα συστατικό ότι υπάρχουν παιδιά με διαφορετικό ε, εθνικό, ιστορικό, δηλαδή προέρχονται από διαφορετικέ χώρε, με διαφορετικέ γλώσσε κτλ. Και όμω ενσωματώνονται σε ομάδε πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας ε, που μόλις κάνατε. Προτείνετε κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα ανθρώπους σαν εσάς και εμάς ε, ε, που ταξιδεύουμε πολύ σε όλη την Ευρώπη. Αν έχει κανείς έναν θεράποντα ιατρό στην πατρίδα του, και χρειαστεί κάτι στις Βρυξέλλες ή κάπου αλλού, δυσκολεύεται να βρει τα αρχαία του. Οπότε η πρότασή σα είναι εξαιρετική. Θα πρέπει να μελετήσουμε να δούμε πώ θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Από την άλλη δεν είναι τόσο απλή όσο θα θεωρούσε κάποιο, διότι φυσικά τα κράτη δεν θα θέλουν να μοιραστούν τι πληροφορίε ε, ούτε να βάλουν τα υπάρχοντα συστήματα τους ε, σε κάτι που δεν γνωρίζουν. Οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε πολλή δουλειά για να τους πείσουμε ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα το οποίο θα είναι πολύ ωφέλιμο για όλους μας. Σίγουρα πολύτιμο αυτό που προτείνετε. Θα πρέπει να το μελετήσουμε. Όσον αφορά την παρουσίασή σας ε, για την παχυσαρκία και τα μέτρα καταπολέμησής της, φυσικά εγώ δεν ήμουν και παλιότερα εδώ στο Κοινοβούλιο όπως κάποιοι άλλοι, ε, ε συγγνώμη, προηγουμένως, οπότε δεν μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ ή κατά του φωτεινού σηματοδότη, αλλά για να συνεχίσω τα όσα είπε η κυρία Κάντεμπαχ, ε, πρέπει να το προσέξουμε. Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο είναι κακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Δεν πιστεύω ότι είναι κακό, εκτό αν πιει κανείς ένα ολόκληρο λίτρο. Ε, αλλά θα ε, σημανθεί με κόκκινο χρώμα λόγω των λιπαρών που περιέχει. Από την άλλη, μια coca Light δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα υγιεινό. Έχει υποκατάστατα ζάχαρη, σπαρτάμι που είναι κάθε άλλο παρά υγιεινή, έχει αποδειχθεί μάλιστα. Αλλά θα επισημανθεί με πράσινο με το σύστημα που προτείνεται. Δεν είναι όμως κάτι που εγώ θα συνέστηνα στους ανθρώπους να το καταναλώνουν, παρότι φυσικά δεν οδηγεί απαραίτητα σε παχυσαρκία. Εμείς στο Λουξεμβούργο προσπαθήσαμε να φορολογήσουμε τη ζάχαρη, την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλλά αυτό θεωρήθηκε λάθος οδό από όλε τι πολιτικέ ομάδε γιατί η καλύτερη λύση είναι να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους, όχι να τους τιμωρούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Στο Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, Coca-Cola, Snickers και τα λοιπά μπορούσε να αγοράσει κανείς ε, μόνο από αυτόματους πολιτές. Και εδώ στην καντίνα πληρώνει κανείς λιγότερο για τις ε, τηγατές του πατάτες παρά για τα ε, λαχανικά του, τα οποία πρέπει να τα ζυγίσει κανείς. Πρέπει να το σκεφτούμε και εδώ στο Κοινοβούλιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά και να δουλέψουμε λίγο και το θέμα της παιδείας. Ευχαριστώ κύριο Στόρβαλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιθανότατα θα έχετε μάθει ήδη δύο πράγματα στη διάρκεια της συζήτησης. Η πολιτική ε, παρότι πρέπει να τηρούν το χρονικό όριο, μιλάνε πολύ. Και από τον συνάδελφο θα ακούσατε, έχει ξεκινήσει ήδη εκστρατεία. Αλλά όταν μιλάμε για την υγεία, ε, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Αν ανοίξω μια φιλανδική εφημερίδα σήμερα, θα βρω ανθρώπους συνομιλικούς μου, οι οποίοι πεθαίνουν και αναγκάζομαι να σκεφτώ για ποιους λόγους. Για, ποιο, για ποιους λόγους ζούμε περισσότερο ή λιγότερο. Ε, το ζήτημα της υγείας μπορεί να είναι κοινωνική, κοινωνικό, μπορεί να είναι θέμα DNA. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι εγώ έχω σχετικά καθαρό μυαλό ακόμα. Περισσότερο σχετίζεται με το DNA της μητέρας μου Πρέπει να μπορούμε δηλαδή να δούμε τα διάφορα ε, ζητήματα με τα οποία σχετίζεται και από τα οποία εξαρτάται η υγεία και να βρούμε τρόπους ε, να παρέχουμε σε ανθρώπους με πιο αδύναμο ή κακό DNA ε, ευκαιρία να ανακαλύπτουν τρόπους ζωής που θα τους βοηθούν στη μακροζωία. Τι να μην τρώνε για παράδειγμα αυτό θα ήταν και ένα τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη ε, ζάχαρη. Όπω ξέρετε, όλε οι μορφέ ζάχαρη δεν είναι κακέ ε, όπω ε, αυτέ που βρίσκει κανεί στα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Χρειάζεται κάποια ποσότητα ζάχαρη για τον καθένα υπό κάποια συγκεκριμένη μορφή. Όταν θα επανέλθουμε μετά από την νίκη μα στι επόμενε εκλογέ, μπορεί να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για σα. Αλλά έχει εξαντληθεί ο χρόνο μου τώρα και θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόρβαλτς και ε, κύριε Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είστε εδώ και για τις εξαιρετικές σας ιδέες. Υπόθηκαν πολλά. Συμφωνά με όσα είπε ο Κριστόφ ε, για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Ναι, φυσικά πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Στη πρώτη προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας. Αλλά υπάρχουν ε, πολιτικές διχογνωμίες δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε, όπως είπε ο Χριστόφ, δεν θέλουμε να ρυθμίζουμε υπερβολικά και να ελέγχουμε υπερβολικά και να λέμε στους νέους ανθρώπους τι να κάνουν. Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να τους λέμε τι να κάνουν. Ίσως να τους προτιμούν και τα κόκκινα ε, από τα πράσινα γιατί τους αρέσουν το απαγορευμένο. Οπότε μην ε, κάνουμε υπερβολική προσπάθεια να απαγορεύουμε πράγματα, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια εκπαίδευση όπως έκανε ο Ομπάμα στη ΣΥΠΑ. Ήταν ο σημαντικότερος πρέσβης ε, ε, τέτοιων θεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, στην εκστρατεία κατά της παχυσαρκίας και έφερε αποτελέσματα με μεγάλη επιτυχία. Οπότε ας ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Αντί να τιμωρούμε και αντί να προσπαθούμε να ελέγχουμε, να δώσουμε κίνητρα και να εκπαιδεύσουμε ε, τους νέους ανθρώπους. Αφορά όλους μας και εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης, η πρώτη σας ιδέα για την ηλεκτρονική υγεία, το συζητήσαμε εδώ χθες, κυρία Πρόεδρε, Έχουμε μια νέα έκθεση για τη διασυνοριακή ε, υγειονομική περιθέλψη και η ηλεκτρονική υγεία είναι μια από τις βασικές πτυχές, από τα βασικά θέματα αυτής της έκθεσης. Μαζί με τον Πέτερ Λίζε και με άλλους εδώ είναι μια από τις βασικές μας φιλοδοξίες ε, να αναπτύξουμε ένα πλήρες αυτόνομο ιατρικό πρόγραμμα στον επόμενο προεπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ηλεκτρονική υγεία θα πρέπει να είναι ένας από του βασικούς πυλώνες, όχι μόνο για την καταπολέμηση της παχυσαρκία, αλλά και για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης του καρκίνου είναι μια κοινή δράση μεταξύ των 27 κρατών μελών ε, στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη και τη επένδυση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Οπότε το πρόγραμμα για την υγεία και ειδικότερα η ηλεκτρονική υγεία θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα όλου αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν πολλά σχόλια για την ιδέα σας και να προσθέσω κάτι. Αν υπάρξει φόρος για ζάχαρη κάπου, ε, το έχετε ψάξει, υπάρχει φόρος για τη ζάχαρη και επιτυγχάνει αποτελέσματα διότι ξέρουμε ότι οι στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση τιμών σε προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη και όχι αύξηση ε, και όχι μείωση απαραίτητα των παχύσαρκων ανθρώπων. Οπότε, τι ήθελα να μας πείτε για την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου φόρου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το σχόλιο σας για το φόρο για την ζάχαρη. Θα απαντήσω τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος ε, μόλις ε, επέβαλε φόρο για τη ζάχαρη. Προς το παρόν ε, έχουμε μείωση των πωλήσεων και αύξηση των τιμών. Και έχετε δίκιο λοιπόν όσον αφορά τα δική μου ομιλία υπάρχει μια παρανόηση και εγώ πιστεύω ότι ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη και ο φόρος για τη ζάχαρη είναι υπεραπλούστευση και ότι χρειαζόμαστε εκστρατείες ε, προγράμματα συγκεκριμένα θετικά, ε, θετικών και όχι αρνητικών κινήτρων στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, πάντα ε, παρατηρείται έλλειψη χρημάτων παντού. Υπάρχουν προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία περιέχουν τόσο πολύ ζάχαρη και είναι τόσο πολύ ενθυγιεινά, με τόσο υπερβολικό τρόπο, που και θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε για να αντλήσουμε κονδύλια για αυτά τα ταμεία. Δεν είμαι λοιπόν εντελώς κατά. Επίσης κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, εγώ έκανα, ε, πρότεινα μια πρώτη ιδέα που συζητήθηκε και στο ΆΗ για τις εξαγωγέ. ώστε ο καθένα μέσω τη Α, συγγνώμη, για τον αθλητισμό και την ε, ένταξη του αθλητισμού της, ε, άσκηση ε, στι επιχειρήσει. Ε, δεν αντέδρασε κανεί σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να αθλούνται περισσότερο καθημερινά. Αυτό θα αποτελούσε μια εξαιρετική εκστρατεία. Διότι πολλέ εκστρατείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται με την παιδική υπαχυσαρκία, αλλά και η υπαχυσαρκία των ενηλίκων είναι επίση ένα θέμα. Για παράδειγμα, όταν εγώ πηγαίνω σε ένα ιατρείο, ε, σε ένα, στο παθολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου. Πολλοί κόσμος έρχεται με προβλήματα στη μέση ε, και η βασική διάγνωση είναι ότι αυτό οφείλεται σε έλλειψη κίνησης. Ε, γιατί να επιβάλλουμε λοιπόν αυτό το φόρο που είπα, γιατί παντού λείπουν τα χρήματα και θέλουμε να χρηματοδοτούσουμε προγράμματα σαν αυτό. Ευχαριστώ. Really Εκτιμάμε ιδιαίτερα τις ιδέες σας. καλό θα ήταν πράγματι να βοηθήσουμε οικονομικά και τις επιχειρήσεις ε, για να εφαρμόσουν ε, την άσκηση στο χώρο εργασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα σας. Βλέπω ότι σε κάποια από τα δικά μας εγχειρήματα έχουμε την υποστήριξή σας και κάποιες από τις δικές σας ιδέες ε, σίγουρα μπορούμε να τις εντάξουμε με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να δούμε πώς. Υπάρχει κάποιο σχόλιο. Να απαντήσω στον κύριο Λίζα, λέει η ομιλήτρια. Στα γερμανικά απάντησε στον κύριο Λίζε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Είμαι Γερμανίδα, έτσι ξεκαθαρίζουμε και το θέμα της εθνικότητας, είναι ίδιο με τη δική σα, Γιατί στη Γερμανία άραγε υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση στο e-health, αλλά και στην τηλεϊατρική και ιδίω από πιο ηλικιωμένου γιατρού είναι αυτό το οποίο ζω και εγώ καθημερινά και νομίζω το πρόβλημα είναι αφενό ότι οι άνθρωποι έχουν πλέον ήδη συνηθίσει στη μεθοδολογία τη εργασία του και δεν έχουν τη θέληση να την αλλάξουν. Από την άλλη μεριά νομίζω επίση ότι οι Γερμανοί ε, ίστανται με πολύ κριτική διάθεση απέναντι σε οτιδήποτε έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα και την ενδεχόμενη έλλειψη προστασίας τους. Θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή η γενιά μας θα αντικαταστήσει τη γενιά των baby boomer και βλέπω εκεί πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό χρήση από πλευρά ιατρών, άλλωστε είμαστε και πολύ πιο κινητικοί από τον παραδοσιακό ε, ε, οικογενειακό ιατρό της παρελθούσας εποχής. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει ήδη να γίνουν επενδύσεις με κάποια προοπτική και υπάρχουν και πολλές πρωτοβουλίες τηλεϊατρικής, ιδίως στον χώρο της Υπέδρου, που έχουν ήδη μεγάλη ε, διάδοση. Γι' αυτό έκανα και την ε, πρόταση αυτή με αυτή την εφαρμογή app η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε σχέση με ένα ε, ε, γενικό, συνολικό ευρωπαϊκό ιατρικό μητρό. Νομίζω θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα έχει το ενδιαφέρον να αναπτύξει ένα μια τέτοια εφαρμογή και ενδεχομένως να επενδύσει σε αυτήν. Θα ήταν πολύ ωραίο λοιπόν να σκέπτεται κανείς προς τα εμπρός, για το μέλλον δηλαδή. Ναι, ευχαριστώ πολύ Βίβια. Ευχαριστούμε. Πρόκειται όντως για ένα θέμα το οποίο αφορά τα, κάτι που και αφορά και μας και τους ε, επόμενες γενιές. Πρόκειται για το... Um, στο θέμα των ε, αποβλήτων και την καταπολέμηση της κατασταπατάλησης των διατροφής και το θέμα, το δεύτερο, είναι το θέμα της χρησιμοποίησης των ε, πλαστικών, κυρίως αυτών που χρησιμοποιούνται μια φορά και που καταλήγουν στα απόβλητα. Λέγεται επίσης ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η χρησιμοποίηση πλαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά και το θέμα επίσης των αποβλήτων. Είναι κάτι που είναι το επόμενο θέμα που θα μας εξηγήσει η Ζουλή Πραντίν. Ευχαριστώ, αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω γαλλικά. Αγαπητοί και αγαπητές ευρωβουλευτές, η πρώτη μου ιδέα είναι ότι υπάρχουν τρία μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει για, κατά τη κατασπατάληση ε, των ειδών διατροφήν ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, η, τα μέτρα αυτά φορούν την αναθεώρηση του θέματος της ημερομηνία λήξης κάποιων τροφίμων, κοινού κανόνες για να μπορεί η διάρκεια συντήρησης κάποιων ειδών διατροφής να γίνεται από κοινού και το θέμα των ε, δωρεών σε είδη διατροφής που πρέπει να κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι ο Διεθνής Οργανισμός που ασχολείται με θέματα ε, γεωργίας και ειδών διατροφής μας λέγει ότι περίπου το 56% των ε, Κατασπατάλησε ήδη ειδών διατροφή, γίνεται από του καταναλωτέ. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθούν κάποια τέτοιου είδου θέματα. Αυτό διότι δεν καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο καταναλωτής ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σημασίας που, αφορ που είναι η ελάχιστη προθεσμία στην οποία πρέπει να καταναλώνονται κάποια είδη διατροφής και ποια είναι τα όρια της κατανάλωσης. Γι' αυτό προτείνω να αλλάξει το θέμα της, ε, των ημερομηνιών που αφορούν τη διάρκεια κατανάλωση των τρυφάνων, να λέγεται δηλαδή κατανάλωση κατά προτίμηση μέχρι και ε, όχι καλό για κατανάλωση μετά. Αυτή είναι μια πρακτική που την έχουν ήδη υιοθετήσει κάποια κράτη όπως η Νορβηγία. Θα πρέπει ε, λοιπόν να ε, χρησιμοποιούνται αυτές οι δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Επίσης, όσον αφορά τις δωρεές που μπορούν να κάνουν σε είδη διατροφής ε, τα σούπερ μάρκετ για είδη διατροφής που δεν χρησιμοποιούνται, να γίνει κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αποτέλεσμα συμφωνία. Όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη καταστραπατάληση των διατροφή, αλλά για να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα τη ε, φτώχεια και τη έλλειψη ειδών διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να μας παρουσιάσετε ίσως και τη δεύτερη ιδέα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η δεύτερη ιδέα μου αφορά τη μείωση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται παντού. Γι' αυτό, αγαπητοί και αγαπητέ ευρωδιαβουλευτέ, ε, θα ήθελα να σα ζητήσω να μπορέσετε να εγκρίνετε τρία μέτρα. Πρώτα απ' όλα, ένα κοινό σύστημα ε, επιστροφής της εγγύησης για τα μπουκάλια που μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής, ώστε να έχουμε την ε, καταγραφή των διαφόρων οικολογικών φορέων και να μπορέσει να υπάρξει φόρους για τις ε, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν και διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των πλαστικών. Ε, βλέπω ότι εσείς εδώ χρησιμοποιείτε δεκάδες πλαστικά μπουκάλια. Θα ήθελα να προτείνω να σταματήσει να ε, παράγονται τέτοιου είδους ε, μπουκάλια που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και να αντικατασταθούν με γυάλινα μπουκάλια. Υπάρχει στη Γερμανία ένα σύστημα επιστροφής εγγύησης. Όταν κάποιος λοιπόν στη Γερμανία αγοράζει ένα μπουκάλι ε, γυάλινο, πληρώνει κάποιο ποσοστό το οποίο του επιστρέφεται όταν γυρίζει γυρίσει πίσω αυτό το μπουκάλι. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε ώστε να έχουμε ένα αηφόρο σύστημα και να αποθαρρύνουμε τη χρησιμοποίηση των πλαστικών στα πλαίσια της οικολογικής και κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να μπορούν τους καταναλωτές για κάποιο τρόπο να τους προωθούμε ώστε να ε, αγοράζουν τα προϊόντα τους με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον. Εγώ πρέπει να σας πω ότι επίσης όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνω πλαστική σακούλα, έχω μια επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα, δεν τρώω κρέας, και ε, παρόλα αυτά υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να αλλάξω. Στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν μπορώ να βρω ε, φρούτα και λαχανικά χίδιν. Τα περισσότερα είναι συσκευασμένα σε μικρά πλαστικά σακουλάκια, πράγμα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό προτείνω να φορολογηθούν και οι διάφορες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλαστικά εκεί που δεν χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε μια κάποια κύρωση όταν χρησιμοποιείται το πλαστικό, όταν μπορεί το προϊόν που πωλείται μέσα στο πλαστικό να μπορέσει να εμφανίζεται διαφορετικά. Και θα πρέπει ο ποιος μολύνει να πληρώνει και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την η φορεία του πλανήτη μας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να αντιδράσουν στις ιδέες σας οι συνάδελφοι, βεβαίως. Θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα αυτό πάρα πολλά πράγματα, διότι οι ιδέες σας επίσης στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας είναι ιδέες που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Όντως, εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στα απόβλητα και στις τόνους πλαστικών, διότι σωστά όπως είπατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ψήφισε μία στρατηγική για την μείωση και σιγά σιγά την μη χρησιμοποίηση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά. Και θέλουμε να διευκολύνουμε τις εναλλακτικέ λύσεις και ξέρουμε ότι Πολλοί μας λένε και το αντίθετο. Αν υπάρχει ανθρακούχο νερό, υπάρχουν κάποια προβλήματα με μια εναλλακτική λύση. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθούν τεχνικέ λύσει για να μπορέσουν να επιληθούν τέτοιου προβλήματα. Μία από τι τροπολογίε μα έγινε υποδεικτή από την Ολομέλεια, δηλαδή να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να μειώνουν κατά 50% την κατανάλωση πλαστικών μία χρήση. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατά πρώτο λόγο απέρριψε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, μετά όμως πέρασε αυτή η τροπολογία στην Ολομέλεια και υπάρχει ε, ένα ε, θέμα ώστε να μπορούν να συγκεντρώνονται κατά 90% τα πλαστικά μπουκάλια. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλους αυτούς τους στόχους Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω, η χρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλας. Αυτή είναι μία κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά τα ποσά και οι αριθμοί στους οποίους καταλήγουμε διαφοροποιούνται πάρα πολύ ανάλογα με ποια χώρα βρίσκεστε. Και ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσεις και να τι χρησιμοποιούμε. Μιλήσατε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής τη Αγγίση. Εγώ είμαι από το Λουξεμβούργο, μια μικρή χώρα, αλλά το υποστηρίζω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα δίκτυα διανομής μεγάλων επιχειρήσεων, όπω η Coca-Cola που έχουν το δικό του δίκαιο ε, δίκτυο συγγνώμη, διανομής. Θα έρθει η Coca-Cola από την Ολλανδία στο Λουξεμβούργο ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Τρίρ της Γερμανίας για να κάνει κάτι, κάτι θα πρέπει να γίνει. Πιστεύω όμως ότι κάνατε μια πάρα πολύ περιγραφή της κατάστασης και τι θα πρέπει να κάνουμε και είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ η κυρία Μπόιλαντ. Δεν νόμιζα θα μου δώσετε ε, τόσο γρήγορα Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια τα οποία γίνανε για τα πλαστικά και να χαιρετήσω τις ε, συνεισφορές που γίνονται. Εγώ ήμουνα και μία από τις ε, ε, εισηγήτριες που αφορούν το θέμα αυτό της χρησιμοποίησης των πλαστικών μία φορά και υπάρχουν θέματα, σκιώδη εισηγήτρια, και υπάρχουν θέματα τα οποία, με τα οποία ασχοληθήκαμε, δηλαδή κυρώσεις ε, που είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το κάνει ε, προσωπικά. Δεν μπορεί όμως έτσι να λύσει το πρόβλημα, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Αυτοί που παράγουν τα πλαστικά θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει να είναι και υπεύθυνοι για το να μας καθαρίζουν από όλα αυτά τα απόβλητα των πλαστικών αυτοί οι οποίοι τα παράγουν. Στο ΕΛΚ, το ΕΛΚ θα πρέπει να το πείσουμε ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει κάποια κύρωση για αυτούς που παράγουν τα ε, πλαστικά. Θα, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω λοιπόν να έρθετε σε επαφή με όσους μπορείτε για να μπορέσουν να επηρεάσουν αυτή την απαγόρευση χρήστης των πλαστικών μίας χρήσης. Επίσης, ε, ε τι άλλο... Ε, σκουπίδι αν θέλετε είναι αυτό το οποίο κατά δεύτερο λόγο ρηπαίνει τις ακτές. Τα ποτσίγαρα. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να δούμε. Τα φίλτρα στα, των τσιγάρων που είναι τα ποτσίγαρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν επίσης να βελτιωθούν. Θα πρέπει όμως να γίνουν ε, κάποια πράγματα και σε επίπεδο κάθε χώρας για την ανακύκλωση. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αλλάξουν τις συνήθειές τους οι άνθρωποι. Διότι μπορεί κανείς να έχει την, χρησιμοποιήσει την πολιτική του μαστιγιού και του καρότου, αλλά αν πρέπει κάποιος ε, να κάνει κάποια χιλιόμετρα για να πάει να ξαναγεμίσει ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι, δεν θα το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι να καταστούν και να αλλάξουν ε, οι βιομηχανίες και σιγά σιγά να πείσουν τον κόσμο να αλλάξει τις συνήθειες με τη δική τους προτροπή πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει γίνει πολλή δουλειά σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάσατε. Όντως, για τα πλαστικά πόβλητα υπάρχει μεγάλη προτεραιότητα σε αυτά που κάνουμε, αλλά Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό από την χρήση των πλαστικών γενικότερα. Τα απόβλητα είναι κάτι διαφορετικά. Επίσης, αν μπορούσε κανείς ε, να χρησιμοποιήσει τα πλαστικά που φτάνουν στα σκουπίδια και να τα ανακυκλώσει, είναι κάτι το διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα μέτρα τα οποία εμείς επιβάλαμε είναι ε, το καπάκι να είναι ε, κολλημένο αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο, να συνδέεται με το μπουκάλι. Uh, Είπαμε λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε. Τώρα όσον αφορά την κατασπατάληση ειδών διατροφής. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο θέμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει πολλή δουλειά για αυτές τις προτάσεις και νομίζω ότι και οι προτάσεις της είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συζητηθεί και συμπεριληφθεί στα διάφορα προτάσεις ψηφισμάτων. Θα δούμε ποιες θα είναι και οι αντιρρήσεις από τα κράτη-μέλη σε αυτό το επίπεδο. Κάποιος άλλος συνάδελφος, η κυρία Κάλεμπαχ ζητά το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και είναι σημαντικό επίσης, ιδίω η νέα, η επόμενη γενέα, η νέα γενέα, να έχει τη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους μας. Θα συνεχίσω από αυτό που είπε η κυρία Βαλεάν. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα διάφορα υλικά, διότι επειδή εδώ εμείς είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, μας ενδιαφέρει λοιπόν και το θέμα των μεταφορών, της μεταφοράς, δηλαδή εκεί όπου χρησιμοποιώ πλαστικά και γυάλινα προϊόντα, είναι και ζήτημα βέβαια βάρους όταν τα προϊόντα αυτά πρόκειται να μεταφορθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Το γυαλί είναι πολύ βαρύτερο από το πλαστικό, συνήθως. Υπάρχουν βέβαια κάποια επιχειρήματα υπέρ, κάποια επιχειρήματα κατά για μεταφορά υγρών, νερού κλπ. για την ε, συσκευασία σε πλαστικές φιάλες δηλαδή. Και είπαμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, για παράδειγμα σε κρίνες, σε ε, σημεία όπου μπορεί κανείς να πάει να προμηθευτεί πρόσιμο νερό, ε, σε παρατίες, σε ε, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ώστε να γίνει πιο ελκυστικό από το να ανοίγει ένα πλαστικό μπουκάλι. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, όλα τα δοχεία, γυάλινα, η πορσελάνινα κλπ. Μετά τη χρήση τους πρέπει να καθαριστούν, πρέπει να απολυμανθούν. Το ζήτημα είναι υπάρχει αρκετό νερό για να, για γίνει αυτή... αυτός ο καθαρισμός. Είναι και ζήτημα υγιεινής. Σκεφτείτε τα νοσοκομεία για παράδειγμα, όπου εκεί είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ε, ε, υλικά συσκευασία μιας χρήσης, ώστε μετά να μπορούν να πετιώνται. Αυτά πρέπει να εξεταστούν στο συνολικό κύκλο του προϊόντος και ποιο προϊόν χρησιμοποιείται σε ποιον τομέα και πώς και γιατί. Δεν μπορεί να είναι κανείς δηλαδή καταρχήν υπέρ ή κατά του πλαστικού. Θα πρέπει να σκεφτεί πόσο επιτυχής είναι η χρήση του κάθε είδους συσκευασίας, ώστε να μην ψηφίζουμε εδώ νομοθετήματα τα οποία ενδεχομένω, αφού θα χρειαστεί για παράδειγμα περισσότερη ε, ενέργεια από ρηκτά καύσιμα για την μεταφορά του βαρύτερου ε, γυαλιού που χρησιμοποιείται για την εμβιάλωση, για την ε, συσκευασία δηλαδή των υγρών και ούτω καθεξής. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτή είναι, ήταν η δική μου παρέμβαση. Σα ευχαριστώ κύριε Κάντενμπαχ. Εσεί τώρα μπορείτε να απαντήσετε εφόσον επιθυμείτε. Just a second. want to add something. Θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο να προσθέσει κάτι. Και εγώ. Ευχώ, θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι. Ο κύριο Χάνσεν. Σε πολλούς τομείς πολιτικής έχουμε σχετικά θέματα. Όπως σήμερα μιλήσαμε το πρωί για τον μηχανισμό γειτονίας, όπου η κυρία Βαριάν ήταν μάλιστα εισηγήτρια ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα και ζητήσαμε 2 δισεκατομμύρια παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις μεταξύ αυτών και την αλλαγή του κλίματος και την αντιμετώπιση των ε, βαρύτατων αρνητικών συνεπειών αλλά και άλλα θέματα όπως η ρήπανση, ρήπανση από πλαστικά ε, θαλασσών και ε, ποταμών. Δεν καταλήξαμε σήμερα σε πλειοψηφία, είχαμε ισοψηφία 26 ε, υπέρ 26 κατά και έτσι χάθηκαν τα 2 δισεκατομμύρια και μία αποχή. Αλλά πρέπει να δούμε σε όλου του τομείς πολιτική τι μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι μονάχα η πολιτική του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Άντσεν. Τώρα εσείς παρακαλώ για να απαντήσετε η εκπρόσωπος των νέων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που το δεν εγκρίθηκε η εκθέση όταν πρόκειται για θέματα περιβάλλοντος και το τι θα βρουν από εμά οι επόμενες γενιές. Το αρνητικό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι όντως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το γιατί χρησιμοποιείται το πλαστικό. Δεν είπα ότι θα πρέπει να απαγορευτούν όλα τα πλαστικά. Ε, είναι ένα υλικό το οποίο πραγματικά έφερε επανάσταση στη ζωή μας. Είναι σημαντικό. Αλλά δύσκολα ανακυκλώνεται επίσης. Γι' αυτό τα μπουκαλάκια Φερρυπίν που συνήθως δεν ανακυκλώνονται με ένα κομμάτι τους, το οποίο δύσκολα επίσης μπορεί να το επεξεργαστεί κανείς για να το ανακυκλώσει. Θα πρέπει λοιπόν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο υλικό στέση των πλαστικών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα και επενδύσει στην έρευνα ώστε α, να χρησιμοποιούν τα ελληνικά. Όντως το κόστος μεταφοράς του πλαστικού είναι χαμηλότερο από το κόστος μεταφοράς του γυαλιού. Αλλά έχουμε να κάνουμε μια πιο οικολογική, ε, ένα πιο οικολογικό υλικό. Χρησιμοποιείται ε, περίπου 50 φορές, ε, δεν κατασκευάζεται από στερεά καύσιμα και ακόμη και αν είναι πιο βαρύ ένα μπουκάλι νερό, είναι καλύτερη συγκεκριμένη περίπτωση να χρησιμοποιείτε το γυάλινο μπουκάλι για το νερό και όχι το πλαστικό. Τώρα, σε σχέση με τις μεθόδους επιστροφής της εγγύησης. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι θα πρέπει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις να, είναι, υπάρχουν όλοι πρόσβαση στο νερό. Ταξίδεψα σε κάποια πόλη σήμερα το καλοκαίρι ε, και εγώ κυκλοφορούσα με το επαναχρησιμοποιούμενο μπουκαλάκι μου, δύσκολα έβρισκα νερό σε πολλές περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το φροντίσει και να το προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβάσιμο νερό παντού. Πόσιμο βεβαίω. Όσον αφορά τα λόμπι, όντως αποτελούν πραγματικό πρόσκομα και θα πρέπει να γίνουν και επενδύσεις σε θέματα παιδείας. Διότι ξέρουμε ότι σε κάθε βιομηχανικό σύστημα Η αγορά είναι αυτή που κανονίζει τους κανόνες. Αν λοιπόν κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις σε θέματα απενδίας και ευνοήσουμε την ε, αγορά ειδών ε, πιο οικολογικών, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και βοηθήσει και την κυκλική οικονομία. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Το τελευταίο μας θέμα είναι η βιώσιμη διαβίωση, ιδέες ε, όπως ε, αστικές ευρύσεις, ε, οροφές, υποδομές, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, προγράμματα καθαρής ενέργειας και σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων, μακροπρόθεσμα. Όλες αυτές οι ιδέες ήταν δημοφιλείς κατά τη συζήτηση στο ΆΙΚΕΣ σήμερα. Έχουμε εδώ την κυρία Άννα Μαρία Ρένερ, η οποία ήρθε να μας παρουσιάσει τις ιδέες ε, των βιώσιμων πόλεων και των οικολογικών ε, τρόπων διαβίωσης. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας ε, και για το ανοιχτό μυαλό που δείχνετε για να ακούσετε τις προτάσεις μας όλες βασίζονται στις καταπληκτικές ιδέες της έκθεσης I. Και χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω κάποιες εδώ αρχικά. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ιδέα μιας Ευρώπης ηγέτιδας στη δημιουργία βιώσιμων συγχρονών πολλών με συστήματα μεταφορών μηδενικών εκπομπών για ανθρώπους και αγαθά, ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε καθαρό αέρα σε όλους τους πολίτες. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιαστεί στην ενδυνάμωση των πρωτευουσών των κρατών μελών. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο. Ενδυνάμωση, χειραφέτηση σημαίνει να παρασχεθούν τα μέσα για να γίνουν πρότυπα πόλεων στις χώρες τους. Ταυτόχρονα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι κάτι απαραίτητο για να ε, οθήσει τους Δήμους προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρότι πολλά οχήματα πρέπει να απογορευτούν στο κέντρο των πόλεων, πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα μεταφορών της πόλης ε, καθαρά μηδενικών εκπομπών με πολύ καλή διασύνδεση ε, και πολύ καλή πρόσβαση σε μικρές αποστάσεις. Ταυτόχρονα η μεταφορά των αγαθών πρέπει να αλλάξει θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο, σε δημοσίες συγκοινωνίες. Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε σημαντικά παραδείγματα ε, μοντέλων χρήσης νέων ενεργειών. Τα βιολεοφορία για, παραδείγματα που χρησιμοποιούνται, για παραδείγμα που χρησιμοποιούνται ε, βάσει βιολογικών αποβλήτων. Χρειάζονται επιχορηγήσει για τι βιολογικέ πόλει, για τι βιώσιμε πόλει, μέσω νέων τεχνολογιών, μέσω προγραμμάτων όπω το, το Ορίζοντα 2020. Αν δούμε για παράδειγμα την πόλη που ζω εγώ, την Αθήνα, είναι μια πολυπληθή ε, πόλη με προβλήματα μόλυνσης. Ε, το να κυκλοφορεί κανεί ω πεζό ε, ή με ποδήλατο είναι επικίνδυνο στην πρωτεύουσα τη Ελλάδα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε οι πόλεις μας να μην εξαρτώνται πια από τα αυτοκίνητα. Στα θέματα της κινητικότητας το ζήτημα είναι ουσιαστικά να παρέχουμε μια ικανοποιητική εναλλακτική στους ανθρώπους. So for the second part, Για το δεύτερο κομμάτι μου ζητήθηκε να μιλήσω για την εκπαίδευση στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δεύτερο πυλώνα για μια καλύτερη Ευρώπη θα ήταν μια Ευρώπη που θα παρέχει κίνητρα στα εκπαιδευτικά τη Ιδρύματα να ηγηθούν τη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πρώτον, χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό των σχολικών προγραμμάτων, νέα σχολικά μαθήματα για την περιβαλλοντική προστασία και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα μπορούσε να προταθεί στι δημόσιε αρχέ των κρατών μελών για την ε, θεωρητική και πρακτική υλοποίηση. Δεύτερον, η Ευρώπη μπορεί να παρέχει οικονομικά και άλλα μέσα στα ε, εκπαιδευτικά της ιδρύματα ώστε να χρησιμοποιούνται χώροι τους ε, για ε, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα σχολεία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα κλείνουν δύο μήνες το καλοκαίρι. Είναι τέλειος χώρος για ηλιακές εγκαταστάσεις που μπορούν να καλύψουν τις ηλεκτρικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως και των γύρω κοινοτήτων και ειδικότερα ε, ε, τα ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται στις ε, διάφορες περιοχές αυτές ώστε να μειωθεί η ενεργειακή ένδυα. Επίσης αυτό μπορεί να παρέχει τεράστιες ευκαιρίες στον τομέα της παραγωγής και της κατανάλωσης. Τρίτον, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τον αριθμό τοπικά οργανικά καλλιεργημένων τροφίμων μέχρι το 2025 προτείνω να υπάρχουν δύο τουλάχιστον υποχρεωτικά πρωινά και μεσημεριανά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια βάσει βιολογικών υλικών και σε άλλα ιδρύματα εκπαιδευτικά. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ε, ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα φρούτα και τα λαχανικά με την οικονομική ε, στήριξη ε, τοπικά παραχθέντων προϊόντων σε όλα τα ιδρύματα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει την περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες της, βελτιώνοντας ό,τι προσφέρουν τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα στον τομέα της περιβαλλοντικής παιδείας. Παιδιά και ενήλικες σε όλη την Ευρώπη μπορούν συστηματικά να μάθουν πώς η κοινωνία μπορεί να ε, μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τη συμπεριφορά μας και τα οικοσυστήματά μας ώστε να ζούμε βιώσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ιδέες σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Γκίζεκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Αναμαρία επίσης για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Προσωπικά ήμουν παρόν και μάλιστα και με επισκέπτες από την Δυτική Κάτω Σαξονία και εγώ και όλοι που συμμετείχαν ενθουσιάστηκαν πολύ από τη συμμετοχή τους στο European Youth Event του Ιουλίου και με ανταλλαγή απόψεων, που στην ουσία ουσιαστικών απόψεων δηλαδή πολύ σημαντικέ, το ζήτημα των βιώσιμων αστικών κέντρων. Γιατί η βιωσιμότητα εδώ συγκεντρώνεται πάντοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγάλη συνένεση. Όλοι είναι υπέρ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, βέβαια, το θέμα είναι πολιτικά θα προτιμήσω απαγορεύσει, επιβολή ποσοστώσεων, αν θέλω την Smart City που προτείνει εσύ, Άννα Μαρία, να περικόψω τόσο πολύ την ατομική μεταφορά ώστε τελικώ να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα, εγώ νομίζω αυτό θα ήταν ο λάθο δρόμο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε πολύ εντατικά το ερώτημα πώ μπορώ να εγγυηθώ τοπικά τον καθαρό αέρα μόνο με χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Διότι μόνο όταν οι εκπομπές που βρωμίζουν τον αέρα μεταφερθούν απλώς λίγα χιλιόμετρα στο στο ε, εργοστάσιο παραγωγή ενέργεια. Βέβαια θα έχει βελτιωθεί ο ατμοσφαιρικό αέρα στην Αθήνα, όμω η μεταφορά, ε, ε όμω η ε, εκπομπή των καυσαερίων, για παράδειγμα του άνθρακα, θα γίνεται κάπου αλλού. Χρειάζεται να αναζητηθούν άλλε δυνατότητε, όπω το car sharing κλπ. Για την εκπαίδευση και διαφώτιση του κοινού, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί είμαι αντίθετο με απαγορεύσει. Έχω τρία παιδιά, 4, 9 και 12 ετών. Και πριν από τα Χριστούγεννα βρισκόμαστε τώρα και όταν δω τι ε, θέλουν ε, ως δώρα, βλέπω καινούριο smartphone, PlayStation, καινούριο computer και λοιπόν αυτά τα πράγματα έχουν άμεση διασύνδεση με κατανάλωση. Έχουμε εδώ Instagram σήμερα για παράδειγμα. συνάδελφοι στέλνουν tweet κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Ε, δηλαδή από τα νέα αυτά μέσα, social media, καταναλώνουν μόνο και περισσότερα. Μίλησες για το Veggie Day προηγουμένως. Έκαναν μια σχετική εκδήλωση κάποιοι συνάδελφοι στην ε, Γερμανία που θεωρήθηκε ως πρόταση για απαγόρευση. Τι κάνουμε λοιπόν με τα νέα μέσα. Μπορείς ε, ας πούμε μαζί με την Veggie Day, δηλαδή την ε, ημέρα χορτοφαγίας, να προωθήσεις και μια μέρα ελεύθερη από smartphone. Θα πετύχεις τότε με μια πέτρα δύο στόχους. Και θα μπορέσεις έτσι ε, να κάνει μια σύσταση στις νεαρές φίλες και νεαρούς φίλους και στους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εσείς και Χάνσιν. Ευχαριστώ πολύ και εσάς Αναμαρία, για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μιλήσατε για το πρόβλημα του επιβαρημένου ατμοσφαιρικού αέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία προσφυγής κατά του Λουξεμβούργου, της ε, πόλης μου, για ε, υψηλά επίπεδα ε, διοξιδίου του άνθρακα. Διότι βέβαια δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένες οι δημόσιες μεταφορές και άλλωστε πολλοί έρχονται και με αυτοκίνητα για να δουλέψουν στην πόλη του Λουξεμβούργου. βλέπετε σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και στο Λουξεμβούργο αλλά και εδώ στι Βρυξέλλε, ένα πρόσωπο μόνο να οδηγεί και να είναι ο μοναδικό επιβάτη δηλαδή. Θα, κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε με το car sharing να επιβαίνουν περισσότεροι στα αυτοκίνητα. Αυτό θα βελτιώσει ήδη πολύ την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Είπατε ότι ζείτε στην Αθήνα. Η Αθήνα βέβαια έχει και ένα μεγάλο λιμάνι και υπάρχει εκεί και ε, μεγάλη κυκλοφορία και φορτηγών πλοίων αλλά και ε, επιβατηγών πλοίων και που φέρνουν πάρα πολύ κόσμο. Και τα μεγάλα αυτά πλοία ε, προκαλούν και σημαντική, και σημαντική ρήπανση. Ακούω για παράδειγμα ότι και στο Βέλγιο, εδώ σε βελικές πόλεις, στην Αμβέρσα για παράδειγμα, συμβαίνει το, σημειώνεται το ίδιο πρόβλημα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ο συναδελφός που μίλησε προηγουμένως τόνισε την ηλεκτρική κινητικότητα. Δηλαδή πράγματι πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, διότι αν αντικαταστήσουμε όλα τα οχήματα με ηλεκτρικά οχήματα και αυτά τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα για παράδειγμα από σταθμούς παραγωγής που καίνε κάρβουνο, τότε δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην πράσινη κινητικότητα. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές και για την ηλεκτρική κινητικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε και πού πρέπει να πάνε να βρούνε όλα αυτά τα ακριβά και σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούν τις μπαταρίες όπως νικέλιο, κοβάλτιο και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και εναλλακτικέ επιλογές που ακόμα όμως δεν υπάρχει επαρκής πολιτική πίεση ώστε να προωθηθούν. Δίνουμε μια προτίμηση στην ηλεκτρική κινητικότητα αλλά παραμελούμε άλλες μορφές ενέργειας. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, να μην έχουμε μια μειοπική αντιμετώπιση δηλαδή του προβλήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας και τις ιδέες που αναπτύξατε βρέθηκα κι εγώ στην Αθήνα και έζησα αυτό το σμόγγ, αλλά ζω και στην Βιέννη και έχουμε παρόμοιες καταστάσεις, όχι τόσο πολύ σμόγγ, αλλά κάθε πρωί έχουμε ε, πάρα πολύ, βαριά κυκλοφορία, πολύ βαριές κυκλοφοριακές εχμές από ανθρώπους που έρχονται με αυτοκίνητα από το περιβάλλον, από τον περίγυρο ας πούμε της ε, πρωτεύουσα. Το ζήτημα είναι πώς αναπτύσσεται παροιμήν και ύπεθρος, ε, πώς διεξάγεται η κινητικότητα στην ύπεθρο, τι προσφέρουμε στο κοινό που ζει εκεί. Εκεί νομίζω η διαθωτική πολιτική και η πολιτική της συνοχής είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα από την πολιτική μεταφορών και την πολιτική περιβάλλοντος. Στην Ήπεθρο, είτε πρόκειται και στην Ελλάδα για παράδειγμα έχετε τα πολλά νησιά, υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης που ίσως να μην καθιστούν αναγκαίο για τους ανθρώπους να πηγαίνουν καθημερινά στην πρωτεύουσα αλλά πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν, εάν και οι βιομηχανίες είναι κατάλληλα ε, εξοπλισμένες, για παράδειγμα, με ευρυζωνικό ε, φάσμα ε, διαδικτύου στην Ήπεθρο. Τα έχουν τα σχολεία τα πράγματα αυτά, τα έχουν τα νοσοκομεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε όταν μιλούμε για κινητικότητα. Και αυτά δηλαδή. Εάν συγκεντρώσουμε την προσοχή μα μονάχα στη βελτίωση τη κατάσταση στα αστικά κέντρα, σημαντικό βεβαίω αυτό και για την, για την ποιότητα τη ζωή, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουμε θεσμού που θα επιτρέπουν στου ανθρώπου όταν θέλουν να εργαστούν, όταν θέλουν να διατηρήσουν ταυτόχρονα τι κοινωνικέ επαφέ του, να είναι δυνατό και να ε, μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα χωρί ε, να αλλάζουν τόπο. Αυτό είναι σημαντικό και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να εξοπλίσουμε ε, την Ήπεθρο, αλλά και απομακρυσμένες περιοχές όπως τα νησιά για παράδειγμα, με τέτοιες συνθήκες διαβίωσης που να καθιστούν, να καθιστούν ελκυστικά για την διαβίωση των ανθρώπων. Βεβαίως, ε, βιώσιμες, τα βιώσιμα αστικά κέντρα έχουν συγκεντρώσει πολύ την προσοχή των Ευρωβουλευτών, έχουμε κάνει πολύ σχετική δουλειά, έχουμε και διάφορα ε, πακέτα για τη στήριξη τέτοιων ιδεών, για smart cities, για ε, βιώσιμες μεταφορές και ούτω Όλα αυτά συμβαδίζουν άλλωστε ως έννοιες. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Μου άρεσε πολύ η ιδέα της ενίσχυσης της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. Αυτό νομίζω πράγματι είναι το πρώτο βήμα Βλέπουμε και ε, την ανάγκη να υπάρξει συνειδητοποίηση και των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών. Όσο περισσότερο συζητούμε για τα πράγματα αυτά, τόσο περισσότερο νομίζω θα ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση και στις χώρες μέλη. Και εμείς είμαστε τελικώς υπεύθυνε για να τα περιλάβουμε αυτά στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θα θέλατε τώρα να απαντήσετε στα σχόλια που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις αντιδράσεις σας. Ε, να τονίσω, έχουμε μόλις 12 χρόνια για να σώσουμε το κλίμα. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Δείτε τη νέα ειδική έκθεση IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Βλέπω στην ατζέντα σας το συζητήσετε χθε. Η έκθεση δείχνει εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα και άλλα ε, αέρια θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν σε όλα ε, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ε, όσον αφορά την κινητικότητα και τις μεταφορές που συζητήθηκαν στο ΆΗ φέτος και γι' αυτό το λόγο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις ιδέες που παρουσίασαν νέοι σε εκείνη την εκδήλωση, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να προβούμε σε τεράστιες αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, μίλησαμε για κάποιες απαγορεύσεις. Η παραγωγή πετρελαιοκίνητων ε, και συμβατικών ε, αυτοκινήτων θα πρέπει να σταματήσει μες στην επόμενη δεκαετία. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέα συστήματα μεταφορών. Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο των 12 ετών είναι τεράστια, αλλά είναι θετική αλλαγή. Αυτό ήθελα να τονίσω εδώ. Όλες οι αλλαγές που θα κάνουμε δημιουργούν για μας ταυτόχρονα και μια καλύτερη ζωή. Μιλάμε μεν για απαγορεύσεις, αλλά η άλλη πλευρά του νομίσματος θα είναι όχι μόνο ο περιορισμός σε 1,5 ε, βαθμό Κελσίου της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και καθαρός αέρας, προστασία των οικοσυστημάτων μας και γενικότερα πιο πράσινα αστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Ήθελα δηλαδή να επικεντρωθώ στα θετικά σημεία των αλλαγών που πρόκειται να κάνουμε όχι να μιλάμε δηλαδή απαραίτητα για απαγορεύσεις και για... Συγγνώμη, έχασα τον ερμό των σκέψεων μου. Ήθελα λοιπόν να τονίσω επίσης ότι όπως είπατε ε, κυρία Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πραγματοποιήσει τεράστιες έρευνες για τις βιώσιμες και έξυπνες πόλεις. Αυτό θα ήθελα να το δω να μεταφράζεται σε γεγονότα. Αν δούμε την Αθήνα αυτή τη στιγμή, ε, κέρδισε το βραβείο κοινοτομία ε, ω πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι γι' αυτό. Διότι έχω δει κάποιε κοινωνικέ και οικονομικέ αλλαγέ, αλλά το κομμάτι τη βιώσιμη ανάπτυξη και του περιβάλλοντο παρα... παραβλέφθηκε εντελώ. Θα ήθελα λοιπόν να δω ταυτόχρονα ένα πιο αυστηρό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και περισσότερη έρευνα. Έχουμε κάνει τόση έρευνα, έχουμε τόσο ε, τεχνολογία, τίποτα φυσικά δεν είναι τέλειο ακόμα. Αφού τα έχουμε όλα αυτά, δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να διστάζουμε να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός. Βήματα που θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγέτιδα στην περιβαλλοντική προστασία. Και εγώ ω Ευρωπαία, ω μισή Ελληνίδα και μισή Γερμανίδα, αυτό θέλω να δω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να δω εμά να ηγούμαστε Τη βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, να δείξουμε στις άλλε χώρες τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ και τα μέλη. Ah, okay. <laughs> yes. um, this was really interesting because I... Αυτό ήταν ενδιαφέρον θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα η μείωση των ζωικών προϊόντων και η απαγόρευση των ορεκτών καυσίμων. Θα έπρεπε ήδη να συζητείτε τώρα. Ωστόσο, προτεραιότητα δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η απαγόρευση ή μια ημέρα χωρίς κινητά τηλέφωνα. Θέλω να εστιαστούμε σε άλλες προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Yeah, well, um, so you never know Πρόεδρος Βαλέαν, Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα βρείτε τις συζητήσεις, ε, τις, μάλλον τις ιδέες που συζητούνται εδώ στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα τη βρείτε σε ψηφίσματα και τελικά στο νομοθετικό έργο. Είναι χρήσιμο λοιπόν να παρακολουθείτε τις εργασίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος που ανταλλάσσει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για το μέλλον των πολιτών και ιδίως για την επόμενη γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στο, στην εκδήλωση και θα σας δούμε στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ.